Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μας υπενθυμίζει ότι η Ένωση βασίζεται στις αδιέρετες παγκόσμιες αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης. Η Ένωση βασίζεται στις αρχές της δημοκρατίας και φυσικά του κράτους δικαίου θέτει τα άτομα στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της, δημιουργώντας ε, την ενωσιακή υπηκότητα και δημιουργώντας μια ευρύτερη, ένα ευρύτερο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Πάνω από οτιδήποτε άλλο, η χάρτα αυτή ε, περιγράφει περί τίνος πρόκειται στην Ευρώπη που θέλουμε και καθορίζει την αποστολή που έχουμε ενώπιόν μας ε, στα θέματα μετανάστευσης και εσωτερικών υποθέσεων. Αντιμετωπίζουμε μια πραγματικότητα στον τομέα αυτό που αποτελεί μεγάλη πρόκληση και σε μεγάλο βαθμό η κοινή μας υπευθυνότητα θα ελέγξει την ταχύτητα της ευρωπαϊκής ενοποίησης και την νομιμοποίηση του ευρωπαϊκού οράματος. Ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα. Το γεωπολιτικό περιβάλλον εκρήγνεται. Έχουμε μια νέα απειλή τρομοκρατίας που έχει δηλώσει ότι προτίθεται να πλήξει τις κοινωνίες μας. Η ευρωπαϊκή οικονομία αγωνίζεται να βγει από την κρίση. Η ήπειρός μας ε, γίνεται όλο και γυρεότερη σε έναν κόσμο που δημογραφικά είναι όλο και νεότερος. Ε, έχουμε γκέτο στις ε, πόλεις μας που αποτελούν το καλύτερο ε, έδαφος για να αναπτυχθούν εξτρεμιστικές ε, ιδεολογίες. Και έχουμε μορφές εγκλήματος πολύ περίπλοκες που δεν γνωρίζουν σύνορα. Και συνεχίζεται η ανθρωπιστική καταστροφή στα σύνορά μας, που είναι οδυνηρή αντίθεση με τις κοινέ ηθικές, πολιτιστικές και πολιτικές αξίες και κληρονομιά μας. Και αντιμετωπίζουμε επίσης την αυξανόμενη έλλειψη ικανοποίησης, δυσαρέσκεια των Ευρωπαίων πολιτών. Θέλω να είμαι σαφής ευθύ εξ αρχή. Η απάντηση στις προκλήσεις αυτές σίγουρα δεν είναι να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη φρούριο. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι τα φρούρια που οικοδομήθηκαν για προστασία από εξωτερικέ απειλές κατέληξαν να είναι φρούρια που έκαναν σκλάβους αυτούς που είχαν στόχο να προστατέψουν και τελικά οδήγησαν σε απομονωτισμό. Μια τέτοια κατεύθυνση δεν είναι τμήμα της εντολής μας. Η Ευρώπη μπορεί να ευημερεί μόνο εφόσον διευκολύνει ενεργά την κινητικότητα των ιδεών, των αγαθών και των προσώπων. Η διαφάνεια και η ασφάλεια είναι πυλώνες ε, του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Αυτή είναι η αποστολή της ε, Επιτροπής σε σχέση με τη μετανάστευση και τις εσωτερικές υποθέσεις. Είναι σαφής αποστολή. Πρέπει η ασφάλεια και η υποβοηθούμενη κινητικότητα να είναι βασικά συστατικά μιας Ευρώπης που θα αναπτύσσεται χωρίς φόβο. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να προστατεύσουμε την ταυτότητα της Ευρώπης ως ένα χώρο στον κόσμο μας που εγγυάται θεμελιώδη δικαιώματα. Πρέπει να εφαρμόσουμε μια ενοποιημένη και στόχο προσιλωμένη πολιτική, ούτω ώστε να προσελκύσουμε το ταλέντο και το εργατικό δυναμικό που χρειάζεται κάθε κράτο μέλο. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα υποστηρίξει την και θα διευκολύνει την ένταξη των μεταναστών στις κοινωνίες μας. Περαιτέρω πρέπει να εγγυηθούμε ότι το έγκλημα και η τρομοκρατία θα αποκλειστούν εκτός των εξωτερικών συνόρων και θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Κυρίες και κύριοι, για τα θέματα μετανάστευσης και εσωτερικών υποθέσεων, εάν δεν κινηθούμε από κοινού ως Ένωση, δεν θα προοδεύσουμε καθόλου. Εάν επιβεβαιωθεί η υποψηφιότητά μου, θα βασιστώ σε εσά, την Επιτροπή Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Πολιτικών Ελευθεριών. Είμαι περήφανος που προτάθηκα ως ο πρώτος επίτροπος για θέματα μετανάστευσης. Αυτό καταδεικνύει τη δέσμευση του, Προεδρε, του Προέδρου Γιούνκερ και της νέας Επιτροπής να αντιμετωπίσουν τις κρίσιμες προκλήσεις της μετανάστευσης. Αντιμετωπίζουμε αυξανόμενο αριθμό ατόμων που επιδιώκουν προστασία εντός των συνόρων μας. Ως Ένωση που δεσμευόμεθα στην τήρηση των ε, παγκοσμίων ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ευθύνη της Ευρώπης να προσφέρει προστασία από τους πρόσφυγες που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και την, ε, τις διώξεις, να σεβαστούμε το δικαίωμα ασύλου και ιδιαίτερα να σεβαστούμε τη ζωή των ε, ανθρωπίνων όντων και το δικαίωμα να μην επαναπροωθούνται σε όλες τις περιστάσεις. Εσείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχετε συμβάλει ουσιοδός στην ε, δημιουργία ενός ρωμαλαίου κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Τώρα έχουμε ένα συνολικό νομικό πλαίσιο και η προτεραιότητά μας θα είναι να διασφαλίσουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν αυτές τις ε, αρχές με ομοιόμορφο τρόπο. Υπάρχουν μερικοί ακόμη συμπληρωματικοί τομείς που πρέπει να συζητηθούν. Ιδιαίτερα η δυνατότητα να οδεύσουμε προς ένα ενιαίο καθεστώς που να ισχύει παντού στην Ένωση βασιζόμενοι και στα αποτελέσματα του ε, ελέγχου του συστήματος του Δουβλίνου θα ε, αναλύσω τα ενδεχόμενα περαιτέρω βήματα. Καθημερινά ακούμε στις ειδήσει ότι φτάνουν και άλλοι μετανάστες στα σύνορά μας και ακούμε απεγνωσμένα άτομα που συχνά ε, ξεκινούν μοιραία ταξίδια στη Μεσόγειο. Ακόμη ένα παράδειγμα τέτοιου προβλήματος είχαμε χθε το βράδυ στην Κύπρο. Πρέπει να αυξήσουμε τη δυνατότητά μας να αντιμετωπίζουμε τις κρίσεις ασύλου, ενώ παράλληλα στηρίζουμε αυτούς, που αντιμετωπίζουν ε, ισχυρές πιέσεις ε, συγκυριακές στα συστήματα ασύλου. χρειάζεται περισσότερη αλληλεγγύη. Και αυτό είναι δυνατό μόνο εάν τα κράτη-μέλη σέβονται και εμπιστεύονται το ένα το άλλο και αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Όμως, ε, Αντιλαμβάνουμε επίσης ότι η πλειονότητα των ε, μεταναστών και αυτών που χρειάζονται διεθνή προσπάθεια βρίσκονται και βρίσκουν καταφύγιο εκτός της Ένωσης από αναπτυσσόμενες χώρες που αντιμετωπίζουν ε, τις δικές τους προκλήσεις. Η διεθνής αλληλεγγύη δεν πρέπει να σταματά στα ενωσιακά σύνορα. Κατά τη γνώμη μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει περισσότερα για να στηρίξει τις χώρες ε, στις περιοχές από τις οποίες προέρχονται πολλοί πρόσφυγες ή από τις χώρες ε, μετάβασης. Θα εργαστώ στενά μαζί με την συνάδελφό μου αντιπρόεδρο Μογκερίνη και τους επιτρόπους που είναι υπεύθυνοι για εξωτερικές υποθέσεις για να δημιουργήσουμε μια περισσότερο συνεκτική πολιτική για τους πρόσφυγες και τη μετανάστευση. Και παράλληλα δεσμεύομαι πλήρως να ενθαρρύνω τα κράτη-μέλη να δεχθούν περισσότερους ε, πρόσφυγες από τρίτες χώρες. Η δυνατότητα μετεγκατάστασης των προσφύγων είναι μία από τις πιο απτές πράξεις ε, γενοδορίας και ελεγγύης έναντι τρίτων χωρών που ε, δίνουν καταφύγιο σε πολύ μεγάλους πληθυσμούς, σε πολύ μεγάλο αριθμό προσφύγων. Η Ένωση πρέπει να προστατεύσει αυτούς που έχουν ανάγκη, αλλά παράλληλα μπορεί να είναι αξιόπιστη αν αντιμετωπίσει την παράνομη μετανάστευση, την παράτυπη μετανάστευση, σεβόμενη πλήρως ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό σημαίνει ότι όσες αιτήσει ε, απορριφθούν πρέπει ε, κατόπιν οι αιτούντες να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και ταχαίως. Η προτεραιότητα πρέπει να είναι να τους βοηθήσουμε να επιστρέψουν εθελουσίως και να τους δώσουμε δυνατότητες να ενταχθούν στις χώρες όπου, ε, από όπου προέρχονται και μάλιστα να ενισχυθούν αυτές τις δυνατότητες επανένταξης. Εδώ πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με τις χώρες προέλευσης, τις χώρες ε, μετάβασης, διέλευσης και ε, επίσης όλους τους διεθνούς, διεθνείς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Μια σφαιρική προσέγγιση φυσικά πρέπει να περιλαμβάνει τη δυνατότητα νόμιμης μετανάστευσης στην Ένωση. Πρέπει να βελτιστοποιήσουμε τα ωφέλη από τη διεθνή κινητικότητα, την μετανάστευση και την ένταξη. Η Ευρώπη είναι τμήμα ενός παγκοσμιοποιημένου και διασυνδεδεμένου πλανήτη, όπου η διεθνής κινητικότητα αναμένεται να αυξηθεί. Πρέπει λοιπόν να αποτιμήσουμε τις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, να εντοπίσουμε τις ελλείψεις που έχουμε σε διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Από πλευράς δεξιότητων η διεθνής ο διεθνή ανταγωνισμό για υψηλού επίπεδου δεξιότητε είναι ήδη έντονο, αλλά η Ευρώπη χρειάζεται επίση εργαζόμενου που θα εργάζονται σε άλλου τομεί. Θέλω να έχω τακτικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ε, τα κράτη-μέλη, τους επιχειρηματίες και τα συνδικάτα. Πιστεύω, μια ευρωπαϊκή ε, πλατφόρμα που να συντονίζει αυτόν τον διάλογο θα ήταν πολύ χρήσιμη. Τα πρώτα έτη εφαρμογής ε, της οδηγίας για την μπλε κάρτα κατέδειξαν, ε, είναι αλήθεια, ότι κατέδειξαν διάφορες ε, αρκετές ελλείψεις. Γι' αυτό ο πρόεδρος Γιούνκερ τόνισε ότι αυτό είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει στην πρώτη φάση των δραστηριοτήτων μας στις πολιτικές του <clears throat> κατευθύνσεις γραμμέ Μία από τις προτεραιότητες μου λοιπόν θα είναι να διασφαλίσουμε ότι οι διαπραγματεύσεις για την οδηγία για τους φοιτητές και ερευνητές θα καταλήξουν το 2015. Και τώρα για το Σέγγεν. Το Σέγγεν είναι τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ενωπήσης και πρέπει να διατηρηθεί η έλλειψη ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Προϋπόθεση για έλλειψη τέτοιων ελέγχων είναι να υπάρχει αποτελεσματικός έλεγχος στα εξωτερικά σύνορα χωρίς, όπως είπα στην αρχή, η Ευρώπη να γίνει φρούριο. Τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο του τμήματος των εξωτερικών συνόρων που τους αναλογεί. Η δυνατότητα της Frontex πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρω για να διασφαλίσουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Όμως τα μέσα που έχουν διάθεσή μας είναι επαρκή. Η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να συζητήσουν, να ξεκινήσουν μια συζήτηση για τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη του Frontex και την ανάγκη και κατά πόσο είναι εφικτό να δημιουργηθεί ένα πραγματικό σύστημα ευρωπαϊκών, ευρωπαίων σύνοριοφυλάκων. Η πίεση στα σύνορα και η λαθρομετανάστευση αυξάνονται συνέχεια. Γι' αυτό πρέπει να αυξήσουμε τη δυνατότητα να αντιδράσουμε για να αντιμετωπίσουμε ολιστικά το πρόβλημα. Ο αποτελεσματικός ε, έλεγχος και διαχείριση των συνόρων πρέπει να βασιστεί στη σύγχρονη τεχνολογία. Πρέπει να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις δυνατότητες που μας προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες για τη διαχείριση της μετανάστευσης και της κινητικότητας. Η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρωπίνων όντων είναι προτεραιότητα. Αυτοί που εκμεταλλεύονται τις ανάγκες των ανθρώπων που είναι σε απόγνωση πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Και η απαράδεκτη μορφή της ε, σύγχρονης δουλείας που είναι η εμπορία ανθρώπων πρέπει επίσης να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά. Είναι λοιπόν κυρίως αυτό μία πάλι εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος και στην Ένωση και διεθνώς και χρειαζόμαστε σφαιρικές απαντήσεις. Οι πολίτες μας ζητούν να τους προστατεύσουμε, καθώς φοβούνται ότι απειλείται η ασφάλειά τους από την τρομοκρατία και τη βία σε καιρούς σειράξεων στη γειτονιά μας και απειλών που προέρχονται από ξένους μαχητές χρειάζεται καλύτερα να αντιμετωπίσουμε και να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα. Το έγκλημα ταξιδεύει ανά την Ευρώπη και υπονομεύει τις κοινωνίες αλλά και τις οικονομίες μας. Χρειαζόμαστε ένα ενημερωμένο πλαίσιο για την ευρωπαϊκή δράση που θα εστιάζει στο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και στις καλύτερες συνέργειες με την εξωτερική δράση η δράση κατά του ηλεκτρονικού εγκλήματος θα διευκολύνει ε, την πλήρη χρήση του διαδικτύου από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Αντίστοιχα, η καταπολέμηση άλλων μορφών οργανωμένου εγκλήματος, όπως το λαθρεμπόριο νοικοτικών, η διαφθορά, θα επιτρέψει ε, στις επιχειρήσεις και στη βιομηχανία να αξιοποιήσουν καλύτερα την εσωτερική αγορά και να αποφευθούν επίσης ε, απώλειες για τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές. Η διατήρηση των δεδομένων είναι ένα μέσο ασφαλείας που έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Τώρα έχουμε ε, την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ε, είναι θέματα προστασίας ε, της δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής και πρόσφατα έχουμε αντιμετωπίσει νέες Απειλέ από τη δρομοκρατία. Ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να βοηθήσει τα κράτη-μέλη στην αντιμετώπιση αυτών των απειλών και ιδιαίτερα τη σοβαρή απειλή των ξένων μαχητών. Θα πρέπει να εργαστούμε ιδιαίτερα στην πρόληψη για την καταπολέμηση ε, της ε, ακραίας ε, ε, αυτής έκφανσης και του εξτρεμισμού. Η συνεργασία της αστυνομίας στην ανταλλαγή προφοριών είναι η ίδια σπονδυλική στήλη της ευρωπαϊκής δράσης στην καταπολέμηση του εγκλήματος και εδώ χωράει πολύ βελτίωση. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχω την πρόθεση να συνεργαστώ στενά μαζί σας έτσι ώστε να έχουμε συγκεκριμένα και αυτά αποτελέσματα. Έτσι ώστε οι πολιτικές στην Ένωση σε θέματα μετανάστευση και εσωτερικών υποθέσεων να στεφτούν με επιτυχία. Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούμε του τομεί όπου η δράση τη Ένωση μπορεί να κάνει τη διαφορά και να βεβαιωθούμε ότι η δράση μα σέβεται απολύτω τα ε, θεμελιώδη δικαιώματα. Αν με επιβεβαιώσετε, θα βοηθήσω τον εκλεγέντα πρόεδρο να χαράξει τι κατευθυντήριες γραμμέ σε θέματα που άμεσα συνδέονται με τη δική μου εντολή σε αυτό το σκοπό θα είμαι σε στενή συνεργασία και μόνιμη επαφή με τον συνάδελφο και αντιπρόεδρο Τίμερ μας και σε αγαστή συνεργασία με τα άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν με επιβεβαιώσετε ε, θα υπηρετήσω και δεσμεύομαι γι' αυτό αυτό που μας ενώνει. Θα σέβομαι ε, με ε, απόλυτη ευλάβεια τις αρχές της Ένωσης, το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και τις αρχές μιας ευρωπαϊκής πολιτικής διαφανούς και δημοκρατικής. Θα είμαι χρήσιμος πολίτης πολίτες χωρίς να είμαι έγκλειστος μέσα σε γραφειοκρατικά τύχη. Ταυτόχρονα θα είμαι αφοσιωμένος στις κοινέ αρχές και αξίες και θα αντιμετωπίζουμε με αποφασιστικότητα και επιμονή ε, τις νέες προκλήσεις. Επίσης, σέβομαι ε, την εντολή που μας έχουν δώσει οι πολίτες. Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι ένας χώρος ελπίδας, προόδου και ελευθερίας υπέρ όλων των πολιτών. Ε, για μένα και για μας είναι ηθική όσο και πολιτική υποχρέωση. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.